Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εθνικοί και ευρωπαίοι βουλευτές, ε, θα ήθελα ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως πρώην Γάλλος βουλευτής να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνεδρίαση για την ε, δημοσιονομική πολιτική και την αποτελεσματικότητα του συντονισμού στον προπολογισμό. Θα συμπροεδρεύσω με τον συνάδελφο Πέτερ Ντούιζενμπερκ, πρόεδρο της Επιτροπής ε, Οικονομικών ε, του Εισβουλής των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών. Να ευχαριστήσω τον Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπο Οικονομικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων, σε θέματα φορολογίας και τελωνίων, που δέχθηκε να κάνει μια ανταλλαγή απόψεων μαζί μας σήμερα το πρωί. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση της Διακυβερνητική συνδιάσκεψης θα συζητήσουμε τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλίσουμε το συντονισμό στα θέματα προπολογισμού και ε, το ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινοβολία. Θα εξετάσουμε τρόπους ε, βελτίωσης, όπως για παράδειγμα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την πιθανή σύσταση ενός μηχανισμού ε, σταθεροποίησης του προπολογισμού για την Ευρωζώνη, όπως αναφέρεται στην έκθεση των πέντε προέδρων με τίτλο «Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης». Αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει οικονομική πολιτική πέραν απλώς της προσθήκης των εθνικών πολιτικών που δεν έχουν συνέργειες μεταξύ νομισματικής πολιτικής και πολιτικής δημοσιονομικής. προτείνεται η δημιουργία ενός προϋπολογισμού της Ένωσης για να καταπολεμήσουμε τα σήματρα σοκ και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορούσε να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό ε, ενός τέτοιου εργαλείου. Θα είναι ουσιαστικά ε, ένας ε, μηχανισμός ο οποίος ε, έχει ένα κεφάλαιο το οποίο ξεκίνησε από συνεισφορά κάθε κράτους μέλους για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες ε, δυνατότητες εγγυήσεων στη συνέχεια είναι σημείο το οποίο δεν ελέγχεται καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου κοινοβουλευτικές έλεγχο. Δεν ελέγχεται ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι σίγουρα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες αν υπήρχε για παράδειγμα ένας υπουργός ε, ε, αρμόδιος ε, για, την, ε, για το Eurogroup, θα είναι υπουργό Οικονομισμών και θα έχουμε και μια διάσκεψη του άρθρου 13 που θα γίνεται ίσως πιο συχνά σε αυτή την περίπτωση, διότι θα εκπροσωπούνται οι Επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικών Θεμάτων των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα έχουμε και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές είναι κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου σίγουρα μας προσφέρει δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσαμε να εξετάσουμε με μεγαλύτερη ε, τόλμη από ό,τι σήμερα. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας ε, και θα περιμένω και τις αντιδράσεις σας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία στη συζήτηση και κατά συνέπεια θα πρέπει λοιπόν να περιοριστείτε στα δύο λεπτά ε, κατά τις παρεμβάσεις σας ή δυνατόν. Ο συνάδελφος Ντούισεμπερκ θα κάνει το συντονισμό και θα δίνει το λόγο στους ομιλητές και στους ε, βουλευτές. Ε, να δώσω καταρχάς ε, το λόγο στον κύριο Μοσκοβισή για μια παρέμβαση το πολύ 10 λεπτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ξεπεράσω τα 10 λεπτά, ελπίζω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για την πρόσκληση εκ νέου, γιατί ήμουν και χθε εδώ για αυτή τη δεύτερη μέρα εργασιών και ανταλλαγής απόψεων. Σήμερα θα εστιάσουμε σε θέματα καθαρά δημοσιονομικά και οικονομικά. Χθες είπα ότι οι προτεραιότητές μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι τριπλά επενδύσεις, διατροτικές αλλαγές και το δημοσιονομικό επί του οποίου θα επικεντρωθώ. Το μήνυμά μου είναι απλό, βεβαίως. Η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι βασικό, βασικό μας μέλημα, αλλά δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη. Και είναι σαφές ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο, ούτω ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και εγώ έχω διατελέσει εθνικός βουλευτής, Βεβαίως όλα τα εθνικά κοινοβούλια λαμβάνουμε πλήρως υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση στα πλαίσια των ευραίων αρμοδιοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων. Ο συντονισμό βεβαίω πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά αναμφισβήτητα ο προσανατολισμός η προσπάθεια να γίνει πολιτικά αποδεκτή η δημοσιονομική πολιτική είναι αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άρα πρέπει να υπάρχει κατανοηση και διάλογος, όπως κάνουμε τώρα. Γιατί είναι τόσο σημαντικός αυτός ο συντονισμός. Για απλό λόγο. Οι οικονομίες, τα χρηματοπιστωτικά πιστήματα των κρατών μελών και ιδιαίτερα της ζώνης ευρώ είναι αδιάρρηκτα δεμένα. Η κρίση μας το δίδαξε ε, με βάση αυτά που μα επέβαλε. Αλλά η κρίση δεν είναι μόνο εσωτερικό θέμα. Συζητήσαμε το θέμα του συντονισμού, αλλά να επενθυμίσω ορισμένα σημεία που θα μα διευκολύνουν, πιστεύω. Πρώτον, η δημοσιονομική ευθύνη είναι πυλώνα ε, των οικονομικών πολιτική τη Ευρώπη. Είναι θεμελιώδη αρχή που πρέπει να συνεχίσει να ισχύει σε αυτήν την μετακρισιακή περίοδο. Είμαι επίτροπος ε, που ασχολούμαι με τα θέματα αυτά και, τον, και τη φορολογία και την ε, τελωνιακή συνεργασία από τον Οκτώβριο του 2015 έχω σαρμοδιότητα αρμοδιότητα ε, να γίνονται σεβαστοί οι δημοσιονομικοί κανόνε. Και πιστεύω ότι αυτή η αρχή της βιωσιμότητα των προπολογισμών δεν είναι μόνο τυπική ευθύνη, είναι πραγματικά ουσιώδης και για την ε, δικαιοσύνη μεταξύ των γενναιών. Να μην ξεχνάμε ότι η Ήπειρός μας ε, θα έχει να αντιμετωπίσει γύρανση του πληθυσμού και άρα ανάλογη αύξηση των δαπανών. Άρα το διακύβευμα είναι να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ του μέσου και βράχη προθέσμου. Μεταξύ της απόλυτης αναγκαιότητας να εξηγιάνουμε τους ε, ισολογισμούς μας, τα δημοσιονομικά μας, αλλά να βοηθήσουμε και την οικονομική ανάκαμψη. Πρέπει να βρούμε σωστές συμβαστικέ λύσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το οποίο συζητήσαμε αναλυτικά χθε. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να κάνουν διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, αλλά πρέπει επίση να βοηθήσουν και την δημοσιονομική βιωσιμότητα μέσω πρόθεσμα. Τελευταίο σημείο που συνδέεται με τον συντονισμό. Η δημοσιονομική ευθύνη σημαίνει να έχουμε μια ενοποιημένη προσέγγιση για την Ευρωζώνη. Σε κάποιε χώρε μπορούν να υπάρξουν ελλείμματα για να γίνουν επενδύσει, αλλά θα πρέπει να διορθωθούν. Σε άλλε χώρε υπάρχουν πολύ περιορισμένε δυνατότητε και υπάρχουν υπερβολικέ προτεραιότητε οι οποίε δεν είναι συνεπεί με τι προτεραιότητε των άλλων κρατών τη Ευρωζώνη. Κάθε φορά πρέπει λοιπόν να διορθώνουμε εκ των προτέρων αυτέ τι ανισορροπίε με μια συνολική προσέγγιση για την Ευρωζώνη συνολικά. Εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε υπερβολικά αναχώρα. Να ορισμένα σημεία κλειδιά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν ασχοληθούμε με το θέμα του δημοσιονομικού συντονισμού. Ξέρετε σε τι πλαίσιο διεξάγονται οι συζητήσεις για αυτόν τον συντονισμό και γενικά για τις ε, δημοσιονομικές ευθύνες. Από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας τα, τα κράτη-μέλη πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές. Το σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη είναι το πλαίσιο για αυτόν τον συντονισμό. Ενώ το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Fiscal Compact στα αγγλικά, είναι διακυβερνητικό και προσπαθεί να ενισχύσει ορισμένες πλευρές αυτού του συντονισμού. Αυτό σημαίνει υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορώ να αρνηθώ ότι η μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνηση που δημιουργήθηκε σε συνθήκε ε, κρίση, το λεγόμενο 2-pack και 6-pack, άλλαξαν τα χρονοδιαγράμματα και μετατόπισαν το κέντρο βάρους της δημοσιονομικής πολιτικής διότι στην Ευρωζώνη τώρα έχουμε ένα μοντέλο συντονισμού εξ άντε των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών δηλαδή το σχέδιο προπολογισμού που υποβάλλεται το φθινόπωρο βασίζεται σε συζητήσεις που έχουν προηγηθεί στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της Ευρωζώνης και ομάδων εργασίας ούτω ώστε να μπορούμε να πούμε και το συζητήσαμε και πρόσφατα για ένα συγκεκριμένο μέλο να μπορούμε να πούμε σε ένα μέλο να επανυποβάλει προπολογισμό. Στην ουσία είναι ένα τρόπο απόρριψη του προσχεδίου προπολογισμού. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι μια ε, σημαντική αρμοδιότητα που έχει κάνει τι δημοσιονομικέ καταστάσει να μεταβληθούν. Οι εθνικέ αρχέ βεβαίω εξακολουθούν να έχουν ένα ρόλο κλειδί. Ιδιαίτερα στα πλαίσια τη ε, δημοσιονομική του ευθύνη. Και είναι τριπλό αυτό ο ρόλο. Πρώτα απ' όλα τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν στη διασφάλιση ο προπολογισμό αυτό να είναι βιώσιμο και να εντάσσεται στα πλαίσια τη ε, Ευρωπαϊκή προοπτική. Υπάρχουν κανόνε. Δεύτερον, έχουν ευθύνη για να είναι αποτελεσματική η δημοσιονομική πολιτική και η πολιτική συνένεση που είναι βάση κάποιου κάθε εθνικού προπολογισμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε βάση μια συζήτηση εθνικής και αποφάσεων για το ποιο θα λάβει τι. Αυτός είναι ο ρόλος ε, που αναμφίβολα πρέπει να παίξει το κάθε εθνικό κοινοβούλιο. Τέλος, τα εθνικά κοινοβούλια είναι οι εγγυητέ της ε, εθνικής αξιοπιστίας στον τομέα των δημοσιονομικών. Ο ρόλος τους είναι οι κυβερνήσει να σέβονται τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει στι Βρυξέλλε. Είναι ισχυρό πολιτικό έλεγχο είναι ένα είδο συνυπευθυνότητα για τα οικονομικά που θα εξελιχθεί περισσότερο στο μέλλον. Τώρα, η συμμετοχή των κοινοβουλίων στου μεσοπρόθεσμου εθνικού δημοσιονομικού προγραμματισμού είναι πολύ σημαντική για τον συντονισμό στα πλαίσια τη Ένωση. Διότι οι εθνικοί αυτοί προγραμματισμοί είναι προπόθεση για τα προγράμματα σταθερότητα και σύγκληση που υποβάλλονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρετε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη απαιτεί κάθε πρόγραμμα να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για το εάν έχει υποβληθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο ο προπολογισμό, αν τον έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, εάν ε, ζητήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου για το προηγούμενο πρόγραμμα ή οποιαδήποτε άλλη σύσταση του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης εφαρμόζουν αυτόν τον οικονομικό συντονισμό στα πλαίσια του, της κατάρτισης των ετησίων εθνικών προπολογισμών στα πλαίσια τη υποβολή του. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν έχουν μια ουσιώδη ευθύνη να εγγυώνται δηλαδή ότι θα λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον καθορισμό των ε, προπολογισμών και των εφαρμοστικών νόμων. Να πω κάτι επίση. Η Κομισιόν, ίσω δεν είναι γνωστό, είναι διατεθειμένη να παρουσιάσει την άποψή τη στα εθνικά κοινοβούλια, αν, επι, είναι κάτι τέτοιο επιθυμητό. Δεν κρυβόμαστε λοιπόν από τα εθνικά κοινοβούλια. Θέλετε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για την αποτίμηση δική μα του προπολογισμού σα, βεβαίω, να κάνουμε αυτό το διάλογο, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Διότι νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετέ ευκαιρίε να μεταβούμε σε εθνικά κοινοβούλια και να κάνουμε αυτή τη ζήτηση σε βάθο, την οποία είναι επιθυμώ. Εάν είναι σημαντικό ο οικονομικό συντονισμό και απαντώ στον Ζαν πρέπει μέσω πρόθεσμα να πάμε και παραπέρα. Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου Γιούγκερ. Εξέφρασε μαζί με άλλους στα πλαίσια τη έκθεση των πέντε Προέδρων και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωση πέρυσι. Ας το πούμε λοιπόν, η ΟΝΕ απαιτεί για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά μία οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική, κοινή ικανότητα. Α το πούμε όπω θέλουμε. Είμαι πεπισμένος εδώ και πολύ καιρό και έχω δεσμευθεί όταν είχα και άλλες ευθύνες επ' αυτού του στόχου. Διότι η κρίση κατέδειξε την έλλειψη κεντρικών δημοσιονομικών φορέων. Ξέρουμε όπως και οι άλλες προηγμένες οικονομίες, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν κάτι τέτοιο. Άρα αυτό θα ήταν μια προϋπόθεση για να υπάρχει ένας προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Και θα μπορούσαμε να έχουμε και ε, ένα Υπουργείο Οικονομικών που θα προσπαθούσε μέσω του προπολογισμού του να ε, ευνοήσει την μακροοικονομική σταθερότητα. Και τέλος, από τη στιγμή που θα υπάρξει προπολογισμό και Υπουργείο Οικονομικών, τότε θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική εκπροσώπηση. Θα πρέπει μια μέρα να υπάρξει ένας υπουργό λοιπόν τη Ευρωζώνη. Θα πρέπει να είναι επίτροπο, θα πρέπει να είναι μέλος του Συμβουλίου, Έχω την άποψή μου και την ε, ε, είχα και παλιά. Και επίσης τα κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό και τα εθνικά πρέπει να οργανώσουν το δημοκρατικό έλεγχο συνεργαζόμενα. Νομίζω ότι οι θέσεις μας είναι πολύ κοντινές ε, κύριε Πρόεδρε και με χαρά να το συζητήσω μαζί σας. Ορίστε λοιπόν μια βασική παρουσίαση. Και τώρα μία απλή παρατήρηση. Βεβαίω, η Κομισιόν είναι βασικός φορέας στον συντονισμό αυτό, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι από, κάτω, από πάνω προς τα κάτω, πρέπει να σεβαστούμε πλήρως την αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτός ο συντονισμός δεν θίγει την κυριαρχία των Εθνικών Κοινοβουλίων και των κρατών. Σας καλώ να κάνουμε πιο συστηματικά αυτό που κάνουμε τώρα να κάνουμε ένα συστηματικό διάλογο για να καταλήγουμε σε κοινέ αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Σίγουρα και η διαρχία για να είναι αποτελεσματική Μερικέ φορές μπορεί να είναι και επιμερισμένη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φραντσέσκο Μπότσι, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, πέντε λεφτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μείνω κι εγώ στο πλαίσιο το οποίο χαράξατε κι εσείς ε, ε, στη σημερινή συζήτηση, ξεκινώντας ε, με μία αξιολόγηση ουσίας. Η Ιταλική νομοθεσία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη στο σύνολο των κανόνων που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει και για τα χρονοδιογράμματα, αλλά και για τον ουσιαστικό σεβασμό των κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσον αφορά το πρώτο, να σας υπενθυμίσω ότι η Ιταλία στην περίοδο που συνέπεσε με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε από το 2008 μέχρι το 2015, βίωσε και χρόνια βαθιών μεταρρυθμίσεων ε, και λογιστικών και προϋπολογισμού μέχρι τη σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο ε, έγινε το Κοινοβουλευτικό Γραφείο Προϋπολογισμού. Αυτό έγινε το 2009 ως μεταρρύθμιση, το 2011 τροποποιήθηκε, το 2012 είχαμε το λεγόμενο ε, ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, που για μας είναι η ισορροπία του προϋπολογισμού και εισήγαγε με μια μεθοδολογία που σήμερα γίνεται αποδεκτή και την εκτιμούν ε, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και στη κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ένα ε, γραφείο του προπολογισμού το οποίο υπερψηφίζεται από τα δύο τρίτα των εκπροσώπων ε, της Βουλής και της Γερουσίας. Όποιος λοιπόν εκπροσωπεί αυτό το όργανο το οποίο εκφράζεται από το, ε, για τον προϋπολογισμό της Ιταλίας έχει εκλεγεί από τα δύο τρίτα της Ιταλικής Βουλής. Πρόκειται για άτομα εγνωσμένου κύρους ε, διεθνούς, αλλά ψηφίζονται, δεν διορίζονται. Και αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς κυρίως ε, και για την αντιπολίτευση, ακόμα και την πιο ακραία αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση για το European Fiscal Council και το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Το Κοινοβούλιο παρεμβαίνει σε όλες τις διαδικασίες και στο προγραμματικό στάδιο και ε, στα ε, ε, θέματα συμφώνου σταθερότητας και προπολογισμού. Και σε ποσοτικό επίπεδο η Ιταλική Βουλή τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις κυρίως για τις μειώσεις και για την καθαρή ε, χρέωση των δημοσίων διοικήσεων. Τώρα, για αυτούς που είναι αντίθετοι στην ε, λιτότητα και αυτοί που υποστηρίζουν ε, τις θεωρίες του Keynes που πολλές φορές τις χρησιμοποιούνται και λαϊκιστές και ευρωσκεπτικιστές για να δικαιολογήσουν την αποτυχία της νομισματικής πολιτικής, ε, δεν αρνούμαστε ότι επειδή υπήρχε μια μακρά κρίση, ιδιαίτερα επαχθής, ε, κυρίως ε, στη μεταπολεμική περίοδο και μετά, και υποχρεώθηκαν πολλές χώρες μέλη να εφαρμόσουν κατά γράμμα ε, τις μεταρρυθμίσεις, ακόμα οι ενδείξεις ανάκαμψης είναι πολύ ισχνές. Αυτό ε, είναι ε, κάτι το οποίο βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό όμω επίση που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η Ευρωζώνη έχει ε, μία πολύ ισχνή αύξηση και σε σχέση με τις αναδεόμενες χώρες αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. και ε, δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε με κάποιες ε, πολυετής συστάσεις. Το λέω πολύ ήπια. Ήταν πολύ σημαντική η κοινωνική κρίση και πολύ δύσκολα μπορούμε να απορροφήσουμε τις συνέπειες σε τόσο σύντομο διάστημα. Ε, χρειάστηκε να εφησιαστούν καταρχάς οι επενδύσεις που αναγκάστηκαν να περιοριστούν κατά πολύ και σε πολλές χώρες μέλες πραγματικά κατέρευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιδράσει, προχώρησε με το σχέδιο Juncker, το οποίο θα έπρεπε να βοηθήσει να υπάρξουν νέες επιπλέον επενδύσεις ε, ε, για 315 δις με 21 δις εγγύησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλή δουλειά επί του σχεδίου Juncker, ε, εμβάθυνε, έγινε εργασία για έξι μήνες, ψήφισε, άκουσε την άποψη όλων και υπέδειξε ένα δρόμο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας δρόμος ίσως λίγο πιο δύσκολος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη εγγύηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε ομόλογα τα οποία θα είναι συμφωνημένα για την ε, ε, χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων. Ε, κάποιοι πιο αισιόδοξοι αναφέρθηκαν σε ευρωομόλογα. Εμείς όμως σκεφτήκαμε κάποια ομόλογα τα οποία θα έπρεπε να έχουν προσυμφωνηθεί για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κοινούς στόχους. Οι μόνες δύο παρεμβάσεις σημαντικών φορέων που βοηθούν είναι το, η ποσοτική χαλάρωση και η σύσταση η οποία ακόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Ταμείου Εξυγίανσης. Και το λεγόμενο European System Mechanism. Τουλάχιστον σε κάποιες χώρες μέλη φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση και ε, ο προπολογισμό δείχνει σημαντικά πλεονεάσματα όχι μόνο στη Γερμανία και στις κατοχώρες, αλλά και στην Ιταλία. Σας το λέω αυτό διότι εάν δεν ίσχυε θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ε, όταν λέω ότι δεν ισχύουν οι εξαγωγές, ε, σας λέω ψε, δεν αρκούν οι εξαγωγές, σας λέω ψέματα. Υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις οποίες δεν πρέπει να υποτιμούμε. Σας το λέω και με αυτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σας το λέω γιατί πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε τις προοπτικές ανάκαμψης της Ευρώπης, όχι μόνο παρεμβαίνοντας όπως έγινε τα τελευταία χρόνια στις εξαγωγές, ε, στην εταιρεία κλείσαμε φέτος με πάνω από 50 δις ε, σε εξαγωγές, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και στην εσωτερική ζήτηση. Και επειδή υπάρχουν και αρκετά άλλα θέματα τα οποία ίσως να ανακύψουν κατά τη συζήτηση, εμείς σε αυτό το τρίμηνο θα ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού της χώρας, προτείνοντας κάποιες καινοτομίε που πηγαίνουν, ελπίζω, προς την κατεύθυνση ε, του συντονισμού που ζήτησε ο Πρόεδρος στην αρχή θα προτείνουμε τη διαγραφή των λεγόμενων ε, σημείων που έχουμε με τις ρήτρες ε, διασφάλισης και θα συντονίσουμε τους μηχανισμούς που συνδέουν τη λειτουργία με το έγγραφο για την οικονομία και τα οικονομικά προς την κατεύθυνση που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης αναφέρθηκε από πολλούς, από υπουργού οικονομικών, ε, τον Επίτροπο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς προσπαθούμε να φανταστούμε ποια μορφή θα μπορούσε να έχει ένας προπολογισμό της Ευρωζώνης. Οι Επιτροπές Οικονομική και η Επιτροπή Προπολογισμών όρισαν δύο εισηγητέ, την κυρία Περβάνου Σεμπερβέση, η Επιτροπή Οικονομικών και τον κύριο Ράιμερ Πόγκε, η Επιτροπή Προπολογισμών για να συντάξουν από κοινού τις προτάσεις τους. Για τρία λεπτά, κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή που αρχίσαμε σήμερα το πρωί είναι ζωτική σημασία. Είναι και μια συζήτηση συγχρόνω που δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας. Να αρχίσουμε τις εργασίες μας με τον κύριο Μπέγκερ και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα έχει αντίκτυπο στην συζήτησή μας και τον προβληματισμό μας και δεύτερον, η νέα πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές οικονομίες μας, κάποιες πρώτα, άλλες αργότερα, σχετικά με την υποδοχή ε, προσφύγων και αυτό το θέμα θα επηρεάσει την ε, συζήτηση που αρχίζουμε βάσει βέβαια των εμπειριών που έχουμε εδώ και χρόνια. Έτσι καλώ το χρονοδιάγραμμα είναι προκαθορισμένο. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει προτάσεις μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα έτσι, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, θα κληθεί να αποφανθεί ρητά για τα ζητήματα αυτά και κάποιες χώρες μέλη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Γερμανία και η Γαλλία όπως θέλετε πείτε το, προβλέπουν επίσης να υποβάλουν πρόταση μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αρχίσει τον προβληματισμό μας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αναγκαστεί να δουλέψουμε με κάπως πρωτότυπο τρόπο, γιατί είναι η πρώτη φορά που έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα της ευκαιρίας ή της δυνατότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει δικό της προϋπολογισμό, που άλλοι δεν το λένε προϋπολογισμό. Επίτα, η Οικονομική Επιτροπή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών επίσης για πρώτη φορά συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Για δεύτερη φορά μάλλον. Η πρώτη φορά ήταν σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο Juncker που ήθελε να εντοπίσει αδυναμίες όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όντως ήταν μια πολύ συγκεκριμένη αδυναμία στην Ευρωζώνη και τώρα μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα με το οποίο οι δύο αυτές επιτροπές συνεργάζονται. Και άλλη μια διευκρίνηση. Το θέμα αυτό πολλές φορές έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήρθε η ώρα να βαθύνουμε περισσότερο. Έχετε μπροστά σας ένα έγγραφο εργασίας το οποίο χτες το βράδυ ολοκληρώσαμε οι δυο μας και που δείχνει με ποιο πνεύμα μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Με έναν ξεκάθαρο στόχο. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση, αλλά από την άλλη μεριά να δουλέψουμε σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως στο έργο και των άλλων θεσμικών οργάνων. Μην αρχίσω τώρα να υπενθυμίζω το ιστορικό του προβληματισμού αυτού. Το μόνο που θέλω να κάνω πριν μου κόψει το λόγο ο πρόεδρος να επιμείνω στο γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί εδώ σήμερα. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη. Αυτό για την Ευρωζώνη σημαίνει ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένας τέτοιος προβληματισμός. Γιατί και τι πρέπει να εξετάσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα σύμμετρα ή συμμετρικά σοκ, πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επενδύσεων και πώς θα διασφαλίσουμε μια πραγματική διακυβέρνηση των οικονομιών μας έτσι ώστε να λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο η Ευρωζώνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, δεν σας έκοψα το λόγο. Ο κύριος Μπέγκε τώρα. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Αυτό το έγγραφο εργασία που εκπονήσαμε από κοινού είναι η αρχή μιας πολύ περίπλοκης διαδικασίας που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μεταξύ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών και Προϋπολογισμών. Αν το κοιτάξετε θα δείτε ότι ασχολείται με το ιστορικό θέμα, με τις προτάσεις των τεσσάρων, την έκθεση των πέντε και με την συμβολή διαφόρων επιστημόνων την οποία θα συμπεριλάβουμε σε ένα περαιτέρω κείμενο και θέτουμε ερωτήματα κυρίως γιατί θέλουμε αυτή η διαδικασία να είναι πολύ ανοιχτή και εσείς ως συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων είστε καλοδεχούμενοι να μας στείλετε εγκαίρως ε, τα σχόλιά σας γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που αποτελεί πρόκληση και που πρέπει από κοινού να το αντιμετωπίσουμε γιατί το θέμα της δημοσιονομικής δυνατότητας της Ένωσης ε, έχει και ένθερμους υποστηρικτές αλλά και αντιπάλους τουλάχιστον ορισμένοι αντέδρασαν αρχικά αρνητικά και ορισμένοι εκφράστηκαν ε, επιφυλακτικά λέγοντας ότι στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας κάτι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε οπότε το θέμα είναι να πούμε ποιος είναι ο κοινός μας στόχος στόχος πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη εδραίωση της ΟΝΕ και οπωσδήποτε τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά. Να μην έχουμε αυταπάτες. Ξέρω ότι η αντιμετώπιση της ε, παρούσης κρίσεως και μάλιστα δεν ήταν μία μόνο η κρίση δεν απλουστεύει τα πράγματα αλλά νομίζω ότι η κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων πρέπει να πάει παράλληλα με την ανάπτυξη προοπτικών που θα μας δείξουν πώς θα διαμορφώσουμε το μέλλον. Αλλά και από αυτού δεν έχω αυταπάτες. Καμία αυταπάτη. χωρίς κοινή και με αλληλεγγύη αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής κρίσης, χωρίς ε, σωστή αντιμετώπιση του θέματος της ε, εγγύησης των καταθέσεων. Εάν δεν αποδείξουμε ότι οι κανόνες που έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό θα εφαρμοστούν πλέον επαρκώς, μια έκθεση για δημοσιονομική ικανότητα γίνεται πολύ δυσχερέστερη. Τραγικά δυσχερέστερη. Γιατί όλα σχετίζονται με όλα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η μακροπρόθεσμη εδραίωση της ΟΝΕ δεν πρέπει να αποκλείει αλλαγές στις συνθήκες. Και η συζήτηση για το τι δυνατότητες θα έχει ο προπολογισμός είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας. Για μένα ορισμένα θέματα είναι πολύ βασικά. Όπως το λέει και η συνθήκη. Ποιος είναι ο στόχος? Μια εσωτερική αγορά που θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς και που θα ευνοεί και θα ενισχύει σε ανταγωνισμό με άλλες υπήρους το δικό μας μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας αγοράς και το νόμισμα το δικό μας είναι το ευρώ και τα υπόλοιπα είναι εξαιρέσεις δηλαδή χώρες οι οποίες αποφάσισαν ε, να μην συμμετάσχουν διαρκώς στο ευρώ δεν θα πρέπει να επιβραδύνουν την πορεία ενοποίησης της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας. Τώρα, εγώ επανειλημμένα ήμουν διαπραγματευτής του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, επειδή δημιουργούμε μια σειρά από επιπλέον ταμεία, με τα οποία συμφώνησε και το Κοινοβούλιο, πρέπει να προσέξουμε να μην θυγεί η ενότητα του προπολογισμού, η ενιαιότητα του προπολογισμού και όταν λέμε ενιαιότητα είναι πραγματικά ενιαίος. Οπότε, τίθεται το θέμα τι δημοσιονομική δυνατότητα θα δημιουργήσουμε, τι διαστάσεις θα έχει και με ποια δομή για τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει όλα αυτά να τα καθορίσουμε. Έλεγχος, ισχυρότερη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού ε, κλάδου ελέγχου γιατί πρέπει να μην επαναλάβουμε το σφάλμα του μηχανισμού σταθερότητας για τον οποίο αποφάσισαν 60 δις τα κράτη-μέλη και στο οποίο συμφωνήσαμε αλλά δεν σέβεται τις ε, δημοσιονομικές αρμοδιότητες ε, των κοινοβουλίων. Βλέπω εδώ τον πρόεδρο Λαμασούρ. Στον επόμενο προβολισμό όμω το διορθώσαμε. Αλλά το γεγονό ότι υπήρχαν 60 δισεκατομμύρια τα οποία μπορούσαν να, τα οποία μπορούσαν να αξιοποιήσουν ε, μέσω του δημοσιονομικού, ε, μέσω των δημοσιονομικών προοπτικών πρέπει πάντα να γίνεται σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση να γίνει πολύ πιο κοινοβουλευτική. Και κάτι ακόμη για τα ταμεία συνοχής. Τα ταμεία συνοχή δημιουργήθηκαν για να οδηγήσουν τις πιο αδύνατες χώρες στην Ευρωζώνη. Άρα, τίθεται το ερώτημα. Αυτές οι χρηματοδοτήσει θα είναι εντό του δημοσιονομικού πλαισίου, θα είναι ειδικοί ή διπόροι και ποιε είναι οι προποθέσει που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να έχουμε τι αναγκαίε πλειοψηφίε για να δημιουργηθούν αυτέ οι δημοσιονομικέ δυνατότητε Και πρέπει να διευκρινίσουμε και τι προσπάθειες πρέπει να κάνουμε εκ των προτέρων στην Ευρωζώνη για να υπάρξει σταθεροποίηση και αξιοπιστία, ούτω ώστε να δώσουμε μια ευκαιρία να είναι ρεαλιστική αυτή η προοπτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπούγκε. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Θα προεδρεύσει ο Πίτερ Ευχαριστώ κύριε Αρτουή. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες σα. Ε, υπάρχουν αρκετά αιτήματα για το λόγο. Θα ήθελα ε, να ακούσουμε τέσσερις ομιλητές πρώτα και να δώσουμε μετά το λόγο στο πάνελ. Αν έχετε ερωτήσεις ως προς το πάνελ, να διευκρινίσετε και σε ποιον ε, την απευθύνετε. Ο κύριος Δίας από την Πορτογαλία. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, για αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα στο δεύτερο πάνελ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις και θα ήθελα να σταθώ σε δύο πτυχές. Η πρώτη είναι η εξής. Έχουμε μια ένωση η οποία βασίζεται στην ειρήνη και στην κοινή ανάπτυξη ο κεντρικός στόχος δεν είναι να υπάρχει σταθερότητα στον προϋπολογισμό. Έχουμε δημιουργήσει πολλά μέσα για να ελέγξουμε και να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια ε, στα δημόσια οικονομικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά λείπουν ακόμα κάποια εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μελών, κυρίως εντός της Ευρωζώνης. Ξέρουμε ότι η δημιουργία προπολογισμού της Ευρωζώνης αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχουμε πραγματικά πολιτική σύγκληση και να μπορέσουμε να επιτύχουμε ή, ε, ε, και να αντιμετωπίσουμε πλήρως ε, τα ασύμετρα σοκ μιας νομισματικής ένωσης που δεν είναι ακόμα η βέλτιστη δυνατή. διάβασα με ενδιαφέρον το έγγραφο το οποίο μας υποβάλλατε και θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη παρατήρηση. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε συνεχώς ε, τη σύσταση σημαντικών μέσων για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια ε, σε επίπεδο επενδυτών, ε, είτε είναι του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και δημοσίου χρέους, τραπεζικά συστήματα και αγορές κεφαλαίων. Διότι η αναβολή αυτή σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες πιέσεις στον εθνικό προϋπολογισμό. Συνεχίζουν να ε, εγγυώνται ε, σε εθνικό επίπεδο οι ε, δημόσιες επενδύσεις και πρέπει να αποτελούν και κίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Κάνω λοιπόν την εξής έκκληση. Η πολιτική προπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να έχει κατά νου ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική σύγκληση. Ευχαριστώ κύριε Τίες. ο κύριος Φαν Άπλτον από την ε, Γερουσία των Κάτω Χωρών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που ανέφερε και ο συνάδελφος Μπάκερ σήμερα από, τη Γαλλική, από την Ολλανδική Γερουσία, που αναφέρθηκε τις, ε, ε, στο πού μπορούν να φτάσουν η διαδικασία απόφασης του δημοσιονομικού συμφένου. Όπως είπε και ένας βουλευτής από την Ιταλία, το σημαντικό ελάττωμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου που δημιουργεί και δημοκρατικό κενό στο ο, θέμα της ε, ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό. Και επομένως πρέπει να υπάρχει ε, και εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας ε, τα οποία στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου αναφέρονται ως ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια. Ο κύριο Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε και σε αυτό σήμερα το πρωί. Εμεί στι κάτω χώρε έχουμε ένα τέτοιο δημοσιονομικό συμβούλιο και πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, μάθουμε και από την εμπειρία μα με αυτό το συμβούλιο. Παρά το γεγονό ότι σεβόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη του, ο ρόλο του στη χάραξη πολιτική στι κάτω χώρε έχει επικριθεί ε, από όλε τι πολιτικέ ε, παρατάξει δίνεται η αίσθηση ότι έχει έναν εξωτερικό ρόλο, διότι η κοινή πολιτική φαίνεται να ε, ε, ε, υπαγορεύεται από πολλά μοντέλα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλο νόημα στην περίπτωση αυτή. Ο, η ενίσχυση του ρόλου αυτών των ανεξάρτητων δημοσιονομικών ε, συμβουλίων ε, μαζί με αυτό το οποίο ζητάτε από την, ε, από την έκθεση των πέντε προέδρων ως επίσημη δημοσιονομική διακυβέρνηση φοβάμαι ότι θα βαθύνει κι άλλο την έλλειψη δημοκρατικής λογοδοσίας Θα ήθελα να θέσω λοιπόν την εξή ερώτηση προς τον κύριο Μοσκοβισή. Πώς βλέπετε εσείς το πρόβλημα αυτό και πώς θα ε, περιορίσουμε περαιτέρω τη δημοκρατική διαδικασία μέσω αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλαν Νίσελη από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μετά τη χρηματοπιστωτική ε, κρίση προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε βασικές προκλήσεις, να μπορέσουμε να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας για να ε, συνεχίσουν τα πράγματα και να αποφύγουμε και μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι σαφές ότι χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποιες πολύ σημαντικές ε, αρχές. Καταρχάς, πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί για τα προβλήματα αυτά στην Ευρώπη και πολύ πιο αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση παντού. Μα ανησυχούν ιδιαίτερα οι συζητήσεις για αυτά τα σχέδια, διότι ε, μου φαίνεται ότι πέραν της αλληλεγγύης χρειάζεται και η προσωπική μας ευθύνη, κυρίως ε, για τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και για τη γενικότερη οικονομική μας πολιτική. Η προσωπική ευθύνη είναι το πρώτο και το κυριότερο, διότι αλλιώς μπορεί να υπάρχει ε, πρόβλημα moral hazard και το έχουμε δει ε, επανειλημμένος αυτό. Μα ανησυχεί το θέμα αυτό, διότι μπορεί να απειλεί και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Επίτροπο Μοσκοβισή πώς βλέπετε εσείς ε, τη λειτουργία του Moral Hazard σε αυτό το πλαίσιο. Thank you. Clear Next Ευχαριστώ, σαφής η ερώτηση. Ο κύριος Μούρεσαν τώρα έχει το λόγο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και βάσει των όσων είπαν οι δύο εισηγητές και κυρίως τον κύριο Μπέγκερ, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που μοιράστηκε μαζί μας το γραφό του. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε στην αρχή της διαδικασίας, γι' αυτό και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ζωτική σημασία. Τώρα, αναφερθήκανε οι επενδύσεις από τον Επίτροπο Μοσχοβησή. Ναι, οι επενδύσεις είναι στοιχείο κλειδί για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη. Θα λέγα όμως ότι το περιθώριο ελιγμών για τις δημόσιες επενδύσεις είναι πολύ περιορισμένο. Οι δημόσιες δαπάνες είναι μεγάλες, σε πολλές χώρες υψηλές. Το περιθώριο ελιγμών είναι λοιπόν πολύ περιορισμένο και το δημόσιο χρέος δεν βοηθάει. Πώς βλέπετε εσείς τον στόχο αυτό για την δημοσιονομική ικανότητα είναι για να οθήσει σε περισσότερες ιδιωτικές ε, επενδύσεις, να μειώσει τις δημόσιες, πώς ε, βλέπετε και τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις δεδομένης ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας, πώς θα γίνουν πιο ελκυστικές οικονομίες μας για ξένες επενδύσεις. Τώρα προς την κυρία Μπέρες για το συντονισμό στην Ευρωζώνη. Ναι, βεβαίως, συντονισμός προς τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες. Άρα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να είναι ο στόχος μας. Θέλω να ζητήσω να προχωρήσουμε σε μια πολύ ειλικρινή τίνη εξέλιξη των εργαλείων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία δαπανώνται μέχρι τώρα, τι γίνεται με τους στόχους μας πώς χρησιμοποιούνται τα οικονομικά εργαλεία αξιολόγησης, ακόμα και τα καινούρια, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις στρατηγικές επενδύσεις, πώς προχωράει. Τέλος, όσον αφορά τη σχέση των χωρών της Ευρωζώνης με εκείνες εκτός. Βέβαια και πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, γι' αυτό και μιλάμε για τη δημοσιονομική ικανότητα. Η αιρεσιμότητα η οποία συνδέεται με αυτή την ικανότητα είναι ζωτική σημασία κατά τη γνώμη μου. Άρα η σχέση μεταξύ χωρών Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης φυσικά πρέπει να ενισχυθεί. Ολοκληρώστε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, δύο κατηγορίες υπάρχουν. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ και πρέπει να τους δώσουμε διασφαλίσεις όπως τον κύριο Κάμερον ότι δεν θα επηρεαστούν από όλα αυτά και υπάρχουν και χώρες που θέλουν και θα μπουν στην Ευρωζώνη κάποια στιγμή μεσοπρόθεσμα μέσα στα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια. Για αυτές τις χώρες πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα αν θέλουν να συμμετέχουν, να δεσμευτούν οικονομικά, να επωφεληθούν, να έχουν δικαίωμα λόγου και να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική ικανότητα να μπορούν να το κάνουν. Ευχαριστούμε. Τώρα, απαντήσεις στις ερωτήσεις. Άκουσα σαφείς ερωτήσεις προς τον κύριο Μοσκοβισή, οπότε θα σας δώσω εσάς πρώτα το λόγο και μετά στους δύο εισηγητές, την κυρία Μπερές και τον κύριο Μπέκη. Πρώτο όμως ο κύριος Μοσκοβισή. Θα ξεκινήσω από την ανάλυση των αναγκών και των ορίων που αντιμετωπίζουμε για να ορίσουμε την οικονομική μας πολιτική και κυρίως τη δημοσιονομική μας πολιτική. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου έχω πει η δημοσιονομική πολιτική τώρα πέρασε από την ύφεση, έγινε ουδέτερη και προχωράει προς την ανάπτυξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η διαδικασία, αλλά έχουν γίνει πολλά στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και εκτός. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις άλλες κρίσεις, το προσφυγικό, την τρομοκρατία, τη δυνατότητα Brexit που ελπίζουμε ότι απομακρύνεται όσο και περισσότερο το θέμα της ελληνικής κρίσης και γενικότερα την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, κοινωνική κρίση και άλλες που απορρέουν από όλα αυτά. Πολύ σοβαρά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε σοβαρή κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λοιπόν μόνο δημοσιονομικές οι κρίσεις. Το σχέδιο Juncker είναι μία προσπάθεια που αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Αντιμετωπίζει την αδυναμία επενδύσεων, την έλλειψη επενδύσεων. Κάτι το οποίο βοηθάει πολύ, αλλά χρειαζόμαστε και δημόσιες πολιτικές που κοστίζουν. Για το προσφυγικό, για παράδειγμα. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόμπλε, μίλησε για την ε, χρηματοδότηση της υποδοχής των προσφύγων. Μίλησε για ένα στάδιο, για ένα πάρος. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει σε αυτό χρησιμοποιώντας κονδύλια. Και δεν πρόκειται για, ένα, ε, κάτι που αφορά τους πάντες. Σίγουρα πρέπει να βάζουμε το σωστό ερώτημα, ότι πρόκειται για μια πρόκληση. Για μια πρόκληση που κρατάει σε χρόνο και που κοστίζει. Και άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να επιδείξουμε αλληλεγγύη και απέναντι στη Γερμανία. Που είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, μεν, αλλά δεν πρέπει να τα αποκριθεί μόνη της σε αυτή την προσφυγική κρίση. Συνεπώς, Υπάρχουν τα όρια της δημοσιονομικής μας πολιτικής και υπάρχουν και οικονομικές ανάγκες. Τρίτον, δημοσιονομική ικανότητα, με δύο λόγια προπολογισμό της Ευρωζώνης. Εδώ πολλά πράγματα πρέπει να αναρωτηθούμε. Πρώτον, να έχουμε ένα τέτοιο προπολογισμό για να το κάνουμε τι. Είδα το εγγραφό σας Υπάρχουν πολλές λειτουργίες που μπορεί να καλύψει ένας τέτοιος προπολογισμό, αλλά δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχει το θέμα της σταθερότητας, υπάρχει το θέμα της ανακατανομής. Όταν ε, μίλησαμε με τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, γιατί και στη Γαλλία συζητιέται πολύ, υπάρχει το θέμα του ελάχιστου επιδόματος ανεργίας. Είναι γενικώ τα επιδόματα, είναι οι επενδύσεις. Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα. Πόσο και θα το μέγεθο του προπολογισμού αυτού και ποιοι θα είναι οι πόροι ενό τέτοιου προπολογισμού. Μην ξεχνάμε και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση Ολόκληρη ότι τίθεται το θέμα των ιδιών πόρων. Ο κύριο Μόντι δουλεύει πάνω σε αυτό. Πάντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε όταν μιλάμε και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό συνολικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα για έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης. Και θα πατήσω στον τελευταίο που πήρε το λόγο, που ρώτησε για τις σχέσεις των χωρών της Ευρωζώνης με εκείνες που είναι εκτός. Προσοχή βέβαια εδώ, γιατί δεν θέλω να κάνω την διασυζήτηση που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όμως, εδώ και τέσσερα χρόνια. Πρώτα ως Υπουργό Οικονομικών και τώρα ως Επίτροπο συμμετέχω και στο Eurogroup και στο ECOFIN. Είναι αναγκαίο να συνεχίζουμε να διαρθρώνουμε καλά τις χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη και εκείνες που είναι εκτός. Παράδειγμα, για την Τραπεζική Ένωση. Συνεργαστήκαμε. Σίγουρα έχει να κάνει με την Ευρωζώνη, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει να έχει αντίκτυπο και στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ήδη λοιπόν υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας. Το ερώτημα είναι πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά στη διάρθρωση αυτή. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάντως αυτό το διτό χαρακτήρα πρέπει να τον σεβαστούμε, να μην τον αμφισβητήσουμε. Βέβαια το ότι υπάρχουν χώρες εκτός Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να εμποδίσει και τις χώρες της Ευρωζώνης να προχωρήσουν περισσότερο. Τέλος για τη δημοκρατία, την υπευθυνότητα, την ηθική. Για να επανέλθω σε αυτά που είπα και στην αρχή, άπαξ και υπάρχει προπολογισμό τη Ευρωζώνη, Υπουργό Οικονομικών, ε, πολιτικέ προ αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει και δημοκρατικό έλεγχο που να βοηθάει στην νομιμότητα, στην νομιμότητα αυτού του θεσμού. Άρα, είπα την πρότασή μου και στους υπουργούς οικονομικών, αν έχουμε προπολογισμό, είναι αναγκαίος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και αυτό είναι που σας εμπλέκει εσάς. Γιατί εδώ τίθενται δύο ζητήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη μια μεριά, το... ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι το Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, αλλά υπάρχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. πώς θα γίνει η διάρθρωση αυτή. Ε, στο φόρουμ αυτό που βρίσκεστε μπορεί κάποια μέρα να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που να γίνει κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Τώρα δεν ξέρω, ο κύριος η κυρια Μπέρες. Παρακαλώ τρία λεπτά ο καθένας. Βεβαίως λέει ο κύριος Μπέγκε. Μια παρατήρηση για αυτά που είπε ο Επίτροπος Μοσκοβισή για το προσφυγικό. Το άρθρο 80 της συνθήκης αναφέρεται σε περίπτωση μαζικών εισρωών προσφύγων για μια σωστή κατανομή των βαρών συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών. Άρα αυτό είναι ήδη εγγεγραμμένο. Αλλά δεν έχουμε εφαρμοστικές διατάξεις και προπολογισμό. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ινστιτούτο για Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές στο Μάνχαεμ έκανε κάποιους υπολογισμούς και λέει ότι η οικονομική διάσταση του προσφυγικού θα μας κοστίσει περίπου 30 δις το χρόνο. 0,2 του ΑΕΠ των κρατών μελών. Εάν γίνει αυτή η χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προοπτικές και τους προπολογισμούς ή να κάνουμε περικοπές από τις δύο βασικές ε, ε, από τους δύο βασικούς λόγους δαπανών που για συγκεκριμένους ε, λόγους θεωρούνται από δύο συγκεκριμένα κράτη-μέλη ιερή και απαραβίαστη. Αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρξει κοινή χρηματοδότηση και να βοηθηθούν οι χώρες που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Αυτό σημαίνει η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η Ελληνική δεν είναι μονόδρομος. Ο κύριος Δίας είπε ότι δεν έχουμε επαρκή όργανα. Βεβαίως πρώτα απ' όλα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα μέσα. Τα διευθυντικά ταμεία πρέπει να βασίζονται περισσότερο στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Βεβαίως αυτό είναι απαραίτητο. Και επίσης τα υπάρχοντα μέσα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικά, κατά πόσο δεν είναι υπερβολικά περίπλοκα κτλ. Κλασικό παράδειγμα η πρωτοβουλία των 6 δις για την αργία των νέων 3 δις νέα, νέο χρήμα 3 δις από το ESF δεν έχουμε μπορέσει να τα εκταμπιεύσουμε όσο θα θέλαμε και θα γιατί μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες νέες δομές για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πιστώσεις πρέπει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μία φράση ακόμη πριν συζητήσουμε για νέο φρέσκο χρήμα προηγείται η καλύτερη νομοθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Α, και εσείς τώρα κύριε Μπότσια μια ερώτηση για τα δημοσιονομικά συμβούλια. Ναι, για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να επαναλάβω μία έννοια την οποία ανέφερα και στην παρέμβασή μου. Είναι προφανές ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Ιταλίας είναι ένα ερετό σώμα και ακριβώς επειδή έχει εκλεγεί τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο και οι αξιολογήσεις που κάνει είναι αξιολογήσεις οι οποίες γίνονται αποδεκτές ομόφωνα. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21 η Οκτωβρίου του 2015 για τη σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου για τα δημόσια ε, οικονομικά με στόχο να συντονίζει τις δραστηριότητες των Εθνικών Δημοσιονομικών Συμβουλίων προβλέπει διορισμούς και αυτό φυσικά είναι εις βάρος της ανεξαρτησίας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητο ένα τόσο σημαντικό συμβουλευτικό όργανο το οποίο συντονίζει τις εργασίες κάποιων ε, εθνικών ε, γραφείων προπολογισμού τα οποία είναι ερετά και όχι ε, με διορισμένους εκπροσώπους. Ε, μία τελευταία παρατήρηση σε αυτό που είπε και ο Επίτροπος Μοσκοβιστή για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Ναι, όπου υπάρχει προπολογισμός υπάρχει και Υπουργό Οικονομικών. Επομένως πρέπει να υπάρξει η λαϊκή βούληση, δηλαδή να έχουμε το θάρρος να βάλουμε κοινά χρέη, ε, κοινέ τραπεζικές εγγύησεις και τον ίδιο Υπουργό Οικονομικών. Δεν θα ξεφύγουμε από αυτό εάν δεν κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα ε, ε, σωστά. Ο φαύλος κύκλος πρέπει να γίνει κύκλος αρετής και πρέπει να σχεδιαστούν όλα αυτά την, ε, ε, και να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Συντομότατα. Χαίρομαι που σε αυτό τον πρώτο γύρο έρωτα απαντήσεων το θέμα των προσφύγων είναι περίπου το πιο σημαντικό γιατί είναι όντως χθες έκανα μία πρόταση πρέπει να αντιμετωπίσουμε θετικά την πρόταση του κυρίου Σόιμπλε που λέει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη σωστή υποδοχή των προσφύγων είναι πολύ ουσιώδες αυτό η Ένωση και ιδίως η Ευρωζώνη πρέπει να δράσουν γιατί αυτή η έκκληση για αλληλεγγύη πρέπει να εισακουστεί όχι μόνο γιατί τίθεται θέμα για τη Γερμανία, αλλά γιατί τίθεται θέμα γενικότερα του τι εννοούμε ως αλληλεγγύη. Ο Πορτογάλος φίλος μας είπε ότι η κατάσταση διαφέρει από κράτος σε κράτος. Μα γι' αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια κοινή θέση για τα δημοσιονομικά αλλά κατόπιν μια ε, προσαρμοσμένη εφαρμογή της. Και τώρα, η δημοκρατική νομιμοποίηση, μην, μα ναι, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συνδιάσκεψη. Αλλά, επιπλέον, εάν έχουμε προϋπολογισμό ευρωζώνης, θα περάσουμε, για παράδειγμα, σε ένα άλλο είδος έμβιου όντω. Δηλαδή αντί να συζητάμε για συντονισμό μεταξύ προπολογισμών, θα συζητάμε για την εφαρμογή ενό προπολογισμού. Άρα θα αλλάξουν και οι σχέσει μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών. Λέτε δεν μπορούν να αυξηθούν συνολικά οι πόροι. Αλλά επειδή δεν θα υπάρξει ανάκαμψη ούτε αμέσω ούτε μακροπρόθεσμα, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη εάν δεν παρέμβει ο δημόσιο τομέα. ακούω να λένε ότι αν υπήρχε μια ενιαία και ιδιαίτερα λειτουργική κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη τότε θα δρούσε ως μαγνήτης για τα κεφάλαια και θα είχαμε ανάκαμψη. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται εγγυήσει του δημοσίου. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά και ελπίζω να καταλήξουμε σε αποτελεσματικές προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε και για τους πολίτες μας τη δυνατότητα του ευρώ να τους χορηγήσει αυτά που δικαίως αναμένουν από ένα λειτουργόν ευρωπαϊκό νόμισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομικών είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε η νομισματική μας ε, ένωση να μην προχωράει με πατερίτσες, αλλά να πατάει γερά στα δυο της πόδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι εθνικές πολιτικές, που μπορεί να είναι πολύ καλές σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να κριθούν ανεπαρκή σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι καλά προσαρμοσμένες σε αυτήν. Το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είχαμε ε, πολιτικές για την μείωση του δημοσίου ελλείμματος, πολύ καλές επίπεδο της κάθε χώρας μέλος, αλλά αν προσθέσουμε όλες αυτές τις πολιτικές, τελικά το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα περιοριστικό και κατέληγε μερικές φορές και στο αντίθετο αποτέλεσμα από την μείωση. Άρα η διακριτική ευχέρεια χρειάζεται, γιατί ο συντονισμός μέσω κανόνων δεν λύνει το πρόβλημα. Η πώληση μίξη, συζήτηση για τις οικονομικές πολιτικές, είναι πράγματα που χρειάζονται. Πρέπει να γίνεται συζήτηση με την κάθε χώρα. Η ιδέα του Πιέρ Μοσκοβισή να πηγαίνει σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και να παρουσιάζει αυτό το πολιτικό μείγμα είναι σημαντικό. Πρέπει να συζητιέται με κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έπειτα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων είναι ζωτική σημασία και για να λύσει τα σύμμετρα σοκ, αλλά και για να επιταχύνει επενδύσεις σε μία περίοδο ύφεση. Για να αποφύγουμε ακριβώς την ύφεση και να αντιστρέψουμε τις τάσεις. Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε επίπεδο της Ευρωζώνης. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφιζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαλαούρας τώρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Perhaps my pronunciation was not correct. Μήπως δεν πρόφερα καλά το όνομα, ρωτάει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπαλαούρας δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Επόμενος ομιλητής, Harvard, από τις κάτω χώρες, τη Δεύτερη Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση και αυτό το τμήμα της έχει να κάνει με τη λύση των προβλημάτων όταν αντιμετωπίζονται αυτά από χώρε από την Ευρώπη και μιλάμε για τη δημοσιονομική ικανότητα. Εγώ θα ήθελα όμως να μιλήσουμε περισσότερο για την πρόληψη του προβλήματος. Και μια αρχή ανεξάρτητη μπορεί να βοηθήσει στο να προληφθούν τέτοια προβλήματα, τα είπε και ο συνάδελφος από τη Γερουσία. Είναι καλό λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει δημιουργήσει το δικό της Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως, το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο Μοσκοβιτζή, είναι κατά πόσο αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι πραγματικά απόλυτα ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτήν. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην περιπλοκότητα των κανόνων, των δημοσιονομικών κανόνων, είτε πρόκειται για τη συμφωνία των έξι οδηγιών, των δύο οδηγιών, είτε πρόκειται για το σύμφωνο σταθερότητας. Όλα αυτά είναι περίπλοκα και οδηγούν σε συζήτηση για την ευελιξία. Επειδή είναι περίπλοκα όλα αυτά, τα κοινοβούλια μας χρειάζονται περισσότερο χώρο για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Μιλήσαμε για το κόστος της προσφυγικής κρίσης. Όντως είναι μια έκτακτη περίπτωση. Αλλά πώς θα πληρωθεί το κόστος. Η αξιοπιστία του συντονισμού έχει να κάνει και με τα μέτρα τα οποία θετούνται. Και εδώ πέρα οδηγούμαστε πολύ συχνά σε έναν αυτοματισμό. Να δεχόμαστε τους προϋπολογισμούς ή να επιτρέπουμε να το κρίνουμε λόγω αμφιβολιών. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σκέτσεφ. Επιτροπή Προϋπολογισμών της Βουλγαρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φυσικά και θα θέλαμε να υποστηρίξουμε όλος ιδιαίτερως την ιδέα εναρμόνισης των δημοσιονομικών πολιτικών και των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών. Χτες συγκεκριμένα συζητήσαμε τη δυνατότητα εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων και ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι η πρώτη προσπάθεια θα είναι η έμεση φορολόγηση να συντονιστεί ίσως να είναι προτιμότερο από το να αναρμονίσουμε την άμεση φορολόγηση. Εκείνος χρησιμοποίησε έναν, μια σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλοποιημένη σύγκριση βέβαια. Όμως η έμεση φόρη όντως είναι διαφορετική στα διάφορες, διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε ρωτάω, τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε αυτήν. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες αν είναι η σωστή. Και έχω και μια άλλη ερώτηση για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι δημοσιονομικά πλεονέσματα έχουμε. Μόνο η Γερμανία είχε τέτοια το 2015 και δεν ήταν αρκετά ούτε καν για να λυθεί το προσφυγικό. Ποιε είναι αυτέ οι χώρε που έχουν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Εγώ δεν βλέπω καμία άλλη εκτό από τη Γερμανία. Πώ λοιπόν θα αποκτήσουμε χρήματα για τον προπολογισμό αυτών που συζητάμε. Αν υπάρχουν άλλα, υπάρχουν πού και πού, μια φορά στα πέντε χρόνια και σε μια-δυο χώρε. Ως εθνικοί βουλευτές εμείς, πώ περιμένετε, για παράδειγμα, να ψηφίσουν οι βουλευτές του Γερμανικού Κοινοβουλίου για να διασφαλίσουν τον προπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου ή κάποιου άλλου. Οπότε η ιστορία αυτή με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Και όταν μιλάμε για τους πρόσφυγες, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες οι χώρες εκείνες οι οποίες ήταν άμεσα εμπλεγμένες στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, γιατί αλληλεγγύη χρειάζεται πάντα και όταν έχουμε προβλήματα. Τώρα η Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι λαμβάνονται δημοσιονομικές αποφάσεις ε, κατά τύχη. Αυτό δεν θα έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό ήδη μου δημιουργεί ανησυχίες. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που τα χρειαζόμαστε για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Ένωσης. Άκουσα πολλά για δημοκρατική νομιμοποίηση σήμερα το πρωί. Αλλά ξέρετε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης υπάρχει άνοδος των εθνικιστικών τάσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη και για τον προπολογισμό και για την οικονομική πολιτική. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουν ότι εργαζόμεθα στους τομείς αυτούς προς το συμφέρον τους. Και ξέρετε, οι πολίτες θέλουν αποτελέσματα, δεν τους ενδιαφέρει η διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Να σεβαστούμε αυτά που αποφασίσαμε στις συνθήκες. Πολλοί αναφέρθηκαν στο Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης. Πρέπει να τηρηθούν όλα, έσουν, όλα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, εάν όλα αυτά έχουν αποφασιστεί με περισσότερη ή λιγότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Του ενδιαφέρει αν όλα όσα αποφασίσαμε είναι τα σωστά διδάγματα από την κρίση. Και γι' αυτό είναι επίσης σημαντικό πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διεύρυνση. Ακούω ότι υπάρχει, συγγνώμη, ε, διεύρυνση, διεύρυνση των οικονομικών μας αρμοδιοτήτων εννοεί ε, ε, ο μιλητής. Βεβαίως, όσο περισσότερο αποφασίζουμε για Υπουργό Οικονομικών, διεύρυνση δημοσιονομικών προοπτικών, τόσο περισσότερο είναι ανάγκη να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη να, ε, ε, αυτά που έχουμε ήδη αποφασίσει. Μόνο έτσι θα αποφασιστούν και θα κρυθούν και ευρύτερε αρμοδιότητε. Η κυρία Πυρέσα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. <clears throat> Αυτά που συζητάμε είναι πολύ σημαντικά. Διότι συζητάμε και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και τη σχέση τους ε, στην προσπάθεια συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ιδιαίτερα για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Γι' αυτό αυτή η συζήτηση είναι περισσότερο πολιτική παρά οικονομική, διότι τα μέτρα τα οποία επιβάλλουν ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά τα τελευταία χρόνια μπορούν να περιγραφούν με μία λέξη. Λιτότητα. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να ζητάτε περισσότερο συντονισμό μόνο και μόνο για να εφαρμόζεται πολιτικές που θίγουν με διαφορετικό τρόπο τις διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, δεν είναι η ίδια επίπτωση της, ε, του συμφώνου για τα δημοσιονομικά στην Πορτογαλία με τη Γαλλία και την Γερμανία. Και οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικές. Είναι επίσης και πολιτικές. Αυτό ήθελα να τονίσω. Διότι, ξέρετε, οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρώπη έχουν σήμερα την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τους βοηθήσει και γι' αυτό είναι εχθρική προς την Ευρώπη ή τουλάχιστον αισθάνονται απογοήτευση. Αυτό οφείλεται στο δημοκρατικό έλλειμμα. Στους περιορισμούς που επιβάλλουν σε ορισμένε χώρες που ποτέ δεν επαρκούν. Πάντα περισσότερες απαιτούνται Οποιαδήποτε χώρα προσπαθεί να κάνει κάτι για του πολίτε τη ισοπεδώνεται. Δεν έχει πια καμία δυνατότητα λήψη αυτονόμων αποφάσεων. Είναι σοβαρό αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, ενώ οι αγορέ κάνουν ό,τι θέλουν για όλου του πολίτε. Εάν μιλάμε λοιπόν για συντονισμό, οικονομικό συντονισμό, πρέπει να μιλήσουμε και για δημοκρατία και για αλληλεγγύη. Και αν μιλήσουμε για δημοκρατία, τότε πρέπει επιτέλους να καταργήσουμε τους μηχανισμού και τους θεσμού που επιβάλλουν τέτοιου. Ε, ε, περιοριστικούς κανόνες ε, στα κράτη-μέλη. Και αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν είναι πραγματικός συντονισμός. Στην ουσία είναι επιβολή από ορισμένε χώρες σε άλλες. Περισσότερο πρέπει να υπάρχει συντονισμός στη δράση μας για τους πρόσφυγες. Και εδώ πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη. Και δεν πρέπει να υπάρχει επιβολή των μεν επί των δε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόι από τη Φιλανδία. Άλλοι δύο μιλητές και μετά θα έχουμε τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Έχουμε λοιπόν πρώτα Φιλανδία και μετά Λετωνία και Γαλλία. Ο κύριο Λόι από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η Ευρωζώνη απαιτεί οικονομικό συντονισμό. Αλλά τώρα που άκουσα τη σημερινή συζήτηση και τις βασικές παρεμβάσεις, ε, ακούω το εξής πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Υπάρχει η πραγματική ε, πραγματικότητα που ξέρουν οι Ευρωπαίοι θύνοντες ε, και αυτοί που ζουν ε, στις χώρες μέλη και μετά υπάρχει άλλη πραγματικότητα, οι πολίτες και τι βιώνουν αυτοί στις χώρες μέλη τους. Αυτές οι δύο διαφορετικές πραγματικότητες δεν θα πρέπει να απέχουν πολύ μεταξύ των. Αλλιώς οποιαδήποτε νομιμοποίηση για τη λήψη αποφάσεων σταματά, αρχίζει να διαβρώνεται. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να υποστηρίξω ένθερμα τις προτάσεις για έναν Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης και τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεν συντονισμός ε, αλλά και την προσωπική ευθύνη των κρατών μελών για τον προϋπολογισμό τους. Ε, θα διαβρωθεί αυτή η προσωπική ευθύνη και λογοδοσία εάν περάσουμε σε ένα κοινό προϋπολογισμό και χρέος. Ο κύριος Πιμιένος από τη Λετωνία. Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πώς ε, σχολιάζετε τις δηλώσεις ότι το επίπεδο λογοδοσίας ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις λογοδοσίας στην ε, Γερουσία των ΗΠΑ δημοσιοποιούνται και μπορεί να τις διαβάσει οποιοδήποτε πολίτης, ενώ σε εμά δεν δημοσιεύονται. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερόμαστε σε πολιτική προπολογισμού και συντονισμό του πολιτι... Ε, προπολογισμού. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να θέσω την ερώτηση στον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, τον κύριο Μοσκοβισή. Η συστημική κρίση στον ε, στεγαστικό τομέα ήταν πολύ σημαντικό ε, θέμα και θα έπρεπε να είμαστε σαφείς. Ήταν υπερβολικό ιδιωτικό χρέος ε, ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων και αυτό ήταν ε, το οποίο οδήγησε στην κρίση και όχι η ε, σπατάλη του δημόσιου τομέα. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Μοσκοβισή να δώσει μια λύση ώστε να μην υπάρχει ενίσχυση του ιδιωτικού χρέους το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα φούσκα. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Λουβαζή από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να αναφερθώ στην κυριαρχία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο κύριε Επίτροπε Μοσκοβισή υπενθυμίσατε το σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών μελών και της κυριαρχίας τους. Θεωρώ ότι αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο και είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ε, πέραν αυτού υπάρχει και ένα στοιχείο σύγκλησης, ε, έτοιμα σύγκλησης σε οικονομικό, κοινωνικό, δημοσιονομικό επίπεδο. Αναφερθήκατε και στις συζητήσεις για την ασφάλιση της ανεργίας και υπάρχει και διάθεση κρατών μελών να καταπολεμήσουν κάποιες μορφές επιθετικών ε, ε, δημοσιονομικών πρακτικών και να υπάρχει και επιθυμία να αποφύγουμε και φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματικότητα που είναι μεταξύ της κυριαρχίας των κρατών μελών και την ανάγκη για σύγκληση. Και θα ήθελα να δω αν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το συνδυασμό. Κυριαρχία των κρατών και σύγκληση σε όλα τα επίπεδα, που είναι το δεύτερο τμήμα του ζεύγους. δεν θα έπρεπε να υποχρεωθούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε ένα από τα στοιχεία αυτή τη σύζευξη. Ε, και υπάρχει και μια κατάσταση ισορροπίας που δεν είναι και τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Και θα ολοκληρώσω την ερώτησή μου λέγοντα ότι ο συντονισμό και η σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλών είναι σίγουρα αποφασιστική σημασία για να καταφέρουμε τελικά να την έχουμε αυτή τη σύζευξη. Ευχαριστώ πολύ. Μία τελευταία αίτηση πριν πάμε στις απαντήσεις ε, και θα ήθελα να προετοιμάσω το πάνελ. Θα έχουν δύο λεπτά το πολύ ο καθένας ώστε να ε, ολοκληρώσουμε πριν από τη μία και τέταρτο. Ο κύριος Καρέλιο από την Ιταλία είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ε, η Επιτροπή θα αποτελείται από ένα πρόεδρο και τέσσερα μέλη, αυτό το Συμβούλιο μάλλον. Το Συμβούλιο αυτό θα αποφασίσει στο μέτρο του δυνατού μέσω συνένεσης, όπως ε, ε, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπου δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση, το Συμβούλιο θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να καθορίσουμε τα προφίλ των μελών του Συμβουλίου αυτού. Και κατά την άποψή μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη με και κάποιες ε, αντικειμενικές πτυχές. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον Επίτροπο Μοσκοβισή είναι ε, η εξή. Με ποιες αντικειμενικές πτυχές ε, θα καθορίσετε τα προφίλ αυτών των ανθρώπων διεθνούς φήμης ώστε το Συμβούλιο να εκπροσωπεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κράτη-μέλη και να γίνονται δεκτές και αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε ως ε, δείγμα την Ιταλική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην επιλογή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και να προσπαθήσετε να έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίου για να καθορίσουμε τουλάχιστον τα αντικειμενικά κριτάρια με τα οποία θα διορίσετε τους, ε, ε, τα μέλη όσο επιτρέπεται με αντικειμενικό τρόπο να διορίσετε αυτά τα μέλη. Κατά την άποψή μας και το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν στην αντικειμενική αξιολόγηση της μεθόδου και των προφίλ. Και μία τελευταία ερώτηση για το ε, καθεστώς και την αποζημίωση των μελών αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει γκρίνει τη σχετική δαπάνη. Ε, έχει υπάρξει κάποιος τίτλος προπολογισμού ο οποίος έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καλύψει αυτά τα περαιτέρω έξοδα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μοσκοβισή για τα τελικά του σχόλια. Δύο λεπτά και δεν θα πω και πολλά πράγματα γιατί είναι σοβαρές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, πρώτη για το μείγμα πολιτικής το μείγμα πολιτικής της Ευρωζώνης σήμερα είναι πιστεύω κατάλληλο και συνδέεται με το θέμα του χρέους που τέθηκε μετά σήμερα θα έλεγα ότι η συμβολή είναι ουδέτερη ή και ελαφρώς θετική για την ανάπτυξη και όπως ξέρετε το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 30% από, την, από το ξέσπασμα της κρίσης και η εξυπηρέτησή του είναι αβάσταχτο βάρος για τις δημόσιες πολιτικές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με πιο συλλογικό τρόπο. Για το χρέος συνολικά, το επίπεδο του δημοσίου χρέους αλλά και του ιδιωτικού είναι θεμελιώδης πρόκληση για την ε, αυριανή μας οικονομική πολιτική. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναέχουμε αυτές τις ε, φούσκες που είχαμε κατά τη δεκαετία 2000. Έχουμε νομίζω πιο ρωμαλαίο τραπεζικό σύστημα. Αλλά το μείγμα πολιτικής πρέπει να αποφύγει. Οτιδήποτε θα θεωρηθεί γύρισμα δηλαδή λιτότητα που θα θίξει την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να αποφύγει και οτιδήποτε θα σήμαινε περιφρόνηση των κανόνων. Διότι τότε θα επανερχόμεθα στις προϋποθέσεις της ε, παρελθούσης κρίσεως. Οι οικονομίες μας ε, ανακάμπτουν, τα συστήματά μας, τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά είναι πιο ρωμαλαία, αλλά όλα εξακολουθούν να είναι ευαίσθητα. Όλοι γνωρίζετε τις πτυτικότητες ε, της παρούσης καταστάσεως. Βεβαίως, είναι δύσκολο να υπάρξουν αποφάσεις με τον κανόνα της ομοφωνίας για τα φορολογικά, αλλά η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι πρέπει να προχωρήσει σε διάφορα θέματα και εδώ χρειάζεται η στήριξη σας. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε φορο αποφυγή, φοροδιαφυγή. Για το θέμα αυτό έχω υποβάλει ένα φιλόδοξο πακέτο που έχει ξεκινήσει να το εξετάζει το Συμβούλιο Κοφίν για τη διαφάνεια με αυτή την ιδέα των αναχώρα εκθέσεων μέχρι πού πρέπει να πάμε. Έχω την άποψή μου, την προσωπική, αλλά πρέπει να κάνω αυτή τη συζήτηση για τον ε, ΦΠΑ την επόμενη εβδομάδα θα το συζητήσει η Κομισιόν αν ε, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό καθεστώς του ΦΠΑ για να αποφύγουμε τις ε, τεράστιες απάτες αλλά βέβαια πολλά θέματα θα παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών εμείς απλώς καθορίζουμε το πλαίσιο δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι η εναρμόνιση αν προκύψει θα προκύψει από τα κράτη-μέλη εμείς θέλουμε να είναι ουσιαστική η φορολόγηση δηλαδή οι πολυεθνικές πρέπει επιτέλους να πληρώσουν εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους, εκεί που προκύπτουν τα κέρδη τους. Και δύο ακόμη για τα δημοσιονομικά συμβούλια. Βεβαίως πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητα. Πρέπει να εκφράζονται εξάντε για την συνολική κατάσταση της Ευρωζώνης και εξ για κάθε χώρα και φυσικά το πώς θα γίνονται οι διορισμοί θα είναι αποφασιστική σημασία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την Κομισιόν στο έργο της. Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρως τις αρμοδιότητές μας για την επιτήρηση του προπολογισμού, αλλά θα μας δώνουν μία αναγκαία συμβουλή και εκεί η ικανότητα και η ανεξαρτησία είναι ουσιώδης. Και για το θέμα της ε, κυρίαρχης απόφασης να υπάρξει σύγκληση. Μα ναι, έτσι κάναμε. Αποφασίσαμε να δημιουργηθεί μια ε, συνένωση εθνικών κυρίαρχων κρατών που προχωρούν με βάση τα στοιχεία που τους ενώνουν. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των ε, Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα τη κοινή προσπάθειά του. Ξέρετε ότι η έκθεση των πέντε προέδρων θέλει να προχωρήσει η ΟΝΕ με πέντε άξονε. Τώρα συζητάμε τον πρώτον, με τι ε, αρχέ των δημοσιονομικών. Η δεύτερη είναι η πιο φιλόδοξη και ουσιαστική, είναι τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία προβλέπετε για τέλος 17. Εγώ ενώπιόν σας είναι να σας καλέσω να μην περιμένετε το 2017 για να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και για να ξεκινήσετε την δημοκρατική συζήτηση που είναι δική σας αρμοδιότητα. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα αυτά των, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Όχι, η συζήτηση για την ΟΝΕ δεν μπορεί να περιμένει μέχρι όλος ο κύκλος πολιτικής να καταλήξει και να έχουμε και το δημοψήφισμα στην ε, Βρετανία και τις εκλογές στη Γαλλία και τη Γερμανία. Η συζήτηση αυτή πρέπει να αρχίσει τώρα. Και με χαρά να συμμετάσχω και εδώ και ενώπιον του κοινοβουλίου σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκε. Ευχαριστώ. Ο Πορτογάλος συνάδελφος η Πορτογαλία συνάδελφος, η Πορτογαλία συνάδελφος είπε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη. βεβαίω. να μην ξεχνάμε ότι έχουμε για το 14 μέχρι το 20 960 δις τα διαρθρωτικά είναι 330 δι, Ανάπτυξη τη υπαίθρου 95 δι, Δηλαδή συνολικά γύρω στα 430 από τα 960 δι, Βοηθάνε τι περιφέρειες. Και τη δική μου περιφέρεια στη Βόρεια Γερμανία. Αυτό είναι έκφραση αλληλεγγύη. Ούτω ώστε για παράδειγμα να εξομοιώνονται οι δυνατότητε ανταγωνιστικότητα να βοηθάμε τις δομές. Ξέρετε, όπως ξέρετε, η φιλανθρωπία αρχίζει από το ίδιο σου το σπίτι. Έτσι ακριβώς το κάνουμε. Τίθεται το θέμα βεβαίως των οικονομικών δυνατοτήτων και των πλεονασμάτων. Στη δική μου χώρα έχουμε το λεγόμενο φρένο χρέους. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Αλλιώς δεν λαμβάνουμε. Ε, δεν κάνουμε αυτό που αρκεί ε, για τη χώρα μας συνολικά. Και σε καλές περιόδους πρέπει να διαχειριζόμαστε του προπολογισμού με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε για τι άσχημε περιόδου και να προκύπτουν ε, δύσκολε καταστάσει. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να συμβάλλει. Αν δείτε το έγγραφο εργασία, ούτω ώστε να διασφαλίζουμε το μέλλον. Τώρα βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε αν το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο ή αν κάτι πρέπει να βελτιώσουμε. Βεβαίω είμαι υπέρ της επικουρικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οικονομική ε, λειτουργία της γιατί μία άκαπτη δομή δεν θα λειτουργούσε. Αλλά βεβαίω, ε, εφόσον ε, καταλήγω εφόσον επιμείνουμε σε πλήρω ανεξάρτητα κράτη και σε απλώς δυνατό συντονισμού δεν θα αντιμετωπίσουμε τις ε, τις ανάγκες ανταγωνιστικότητας. Η κυρία Μπερές, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, πολύτιμη για τον κύριο Μπέγκε και για μένα. Είπα και πριν ότι έχετε μπροστά σας κάποια έγγραφα που μόλις βγήκαν φρέσκα φρέσκα και είπα ότι είναι προνόμιο αυτό για σας. Σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο σε όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καλό να μπορέσουμε όλοι μαζί να ορίσουμε το πλαίσιο δημοκρατικής νομιμότητας μέσα στο οποίο θα προχωρήσουμε για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Σίγουρα είναι βαρύ το καθήκον. Το είπα και το αναφέρω και στο έγγραφο εργασία. Και το ξέρω ήδη από την εποχή των εργασιών του Μακντάγκαλ το, τη δεκαετία του 70 αλλά πρέπει βέβαια να τα ξαναδούμε όλα αυτά βάσει των κρίσεων που αντιμετώπισε η Ευρωζώνη και βάσει των όσων ζούμε σήμερα. Το είπαμε αυτό, είπαμε ότι είναι αναγκαία η αλληλεγγύη για την υποδοχή των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Τέλος ο κύριος Μπότσια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνοντας ε, με κάποιες από τις παρενέσεις που ε, μας έγιναν. Να υπενθυμίσω ότι όλοι έχουμε δύο πολύ σημαντικά ε, ραντεβού. Το ένα είναι η επικαιροποίηση της στρατηγικής 2020, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αναγνώριση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, αλλά επίσης και των όσων δεν έχουν ε, λειτουργήσει. Ε, υπήρχαν απογοητευτικά αποτελέσματα όσον αφορά το στόχο της αύξησης της απασχόλησης και τη μείωση της ένδειας η προοπτική της ενσωμάτωσης του Δημοσιονομικού ε, Συμβουλίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας νομίζω ότι θα μπορέσει να αποτελεί σοβαρή ε, επίπτωση στα μακροοικονομικά ζητήματα και στα δημοσιονομικά ζητήματα. Αυτές οι δύο συναντήσεις που μας αφορούν όλους ε, είναι ένας τρόπος να επαληθεύσουμε αν πρέπει να γίνει κάποια περαιτέρω διόρθωση στους εφιστάμενους κανόνες, ε, ξεκινώντας από την ε, συνολική εφαρμογή των κείμενων κανόνων που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή για όλες τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε τα όσα προέκυψαν από την ε, ανάδυση ε, ολόκληρων και αυξανόμενων πλεονασμάτων, όχι μόνο στις εξαγωγές, αλλά και των ε, δημοσίων προπολογισμών. Ευχαριστώ. Πριν δώσω τελικά το λόγο στον κύριο Αρτουή για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση, ένα σχόλιο για τα διαδικαστική. Θα ξεκινήσουμε στις 3 παρατέταρτο. Ε, έχουμε λοιπόν ένα τέταρτο επιπλέον για το διάλειμμα. Κύριε Αρτουή, ευχαριστώ να φτάσουμε λοιπόν στα συμπεράσματα. Χαίρομαι για την ε, σημερινή συζήτηση. Ήταν μια πλούσια συζήτηση. Και εν τέλει αναλάβαμε ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο όταν αποφασίσαμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νόμισμα, το ευρώ. Ε, φτιάξαμε ένα νόμισμα ορφανό από χώρα και ε, προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με τον καθορισμό ενός κανονισμού συνειδιοκτησίας, δηλαδή μέσω κανόνων. Διαπιστώσαμε όμως ότι δεν είμαστε σε θέση να ε, γίνουν σεβαστές οι παραβιάσεις και να τις τιμωρήσουμε τις παραβιάσεις και εκεί αποδείχθηκαν τα όρια του νομίσματος όταν αντιμετωπίσαμε την ελληνική κρίση. Και νομίζω ότι το επίπεδο ε, ανάπτυξης σε όλη την Ευρωζώνη ε, δεν ε, είναι τόσο ικανοποιητικό. Υπάρχει πολύ σημαντική ανεργία σε αρκετές χώρες και μας ενδιαφέρει και η σωστή διακυβέρνηση. Νομίζω ότι η Ευρωζώνη έχει μια ιδιαίτερη αλληλεγγύη όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό ε, σταθερότητας. Ε, δεν συμμετείχαν εκεί οι 28, συμμετείχαν τα μέλη της Ευρωζώνης. Και αυτή η αλληλεγγύη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση. Και το είπαμε άλλωστε, σαφώς και υπάρχει μια απόπειρα να υπάρχει ένα μείγμα πολιτικής, αλλά υπάρχουν και κάποια ε, σημαντικά στοιχεία προόδου. Ε, πιστεύω ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί ε, να γίνει πιο ισχυρή μέσω της σύστασης μιας ομάδας εποπτείας στην οποία θα συμμετέχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου μας προσφέρει ε, τεράστιες δυνατότητες να το επιτύχουμε αυτό. Όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωζώνης, κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία γιατί υπάρχει μια έκθεση εν εξελίξη και ε, πρέπει να σας πω ότι πρέπει κατεπηγόντως να προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό ε, θα πρέπει να δείξουμε και κάποια τόρμη εδώ και αν ε, κρίνω από την κοινή γνώμη νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους ε, ενδιαφέρονται για το ευρώ και οι Ευρωπαίοι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωζώνης περιμένουν μια ουσιαστική βελτίωση της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Ε, ας προσπαθήσουμε να μην τους απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστώ.